γίνει το ψήφισμα πιο συμπαγές και αφού βρούμε συμφωνία θα ανατρέξουμε το κείμενο, θα το κάνουμε πιο ευανάγνωστο και αποτελεσματικό όσο γίνεται. Ώστε είναι κάτι, να είναι κάτι το χαρμόσυνο σαν το στενιάδικο δέντρο λέω μιλήτρια. Τώρα βέβαια για τις διάφορες χώρες ε, δεν είμαι κατά να αναφερθούν αν είναι σαφείς οι αναφορές και να μην καταλήξουμε σε ένα κατάλογο τέλο πάντων μια παρήθμιση παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού στον κόσμο. Αλλά να αναφέρεται τέλο πάντων μια σαφή στάση τάση που αφορά τέλο πάντων νομοθεσίε που αραβιάζουν ανθρώπινα δικαιώματα ή κάτι παρόμοιε καταστάσει. Αυτό νομίζω αξίζει να το πούμε. Είναι καλή λοιπόν η διαδικασία που ακολουθούμε και σήμερα μας υπενθυμίζονται οι δικές μας ευθύνες και η ανάγκη για ευρωπαϊκή ηγεσία παγκοσμίω και πρωτοπορία η οποία είναι περισσότερη επίκαιρη από ποτέ. Ναι, ευχαριστώ για τους πράσινους Μπαρα Λοχμίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εμείς στην ομάδα είμαστε ικανοποιημένοι με την έκθεση και ελπίζουμε ότι θα έχουμε και καλά αποτελέσματα στην ψηφοφορία. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, γιατί ήμασταν ε, πολύ αποτελεσματικοί, όχι πολύ γρήγοροι, αλλά συγκεκριμένοι και συμπαγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ε, όποιος μας ακούσει προσεκτικά, όποιος διαβάσει αυτή την έκθεση, όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, θα δει ότι έχουμε στην Ευρώπη, εδώ στις χώρες μας, μια κοινωνία των πολιτών και ανθρώπινα δικαιώματα που ε, έχει μια μικρή διαφοροποίηση και αυτό το συζητάμε κάθε χρόνο και το διαβάζουμε στις εκθέσεις ε, και με τους, το συζητούμε και με τις συγκεκριμένες μη κυβερνητικέ οργανώσεις που εμπλέκονται. Ε, είχαμε μια πολύ καλή βέβαια βάση επικοινωνίας με, μεταξύ μας, αλλά σε αυτή την περίπτωση με την Κομισιόν δεν υπήρχε αυτό δεν πρέπει μόνο μερός να αποφασίζει το εξή ε, να αντιδρά γραπτός στις εκθέσεις μας. Μπορεί να έχουμε χιλιάδες ε, τροπολογίες συμβιβαστικές, αλλά όταν γίνεται γραπτή απάντηση σε βουλευτές που κάπου διαφωνούν, καταλαβαίνετε. Τώρα, υπάρχει το θέμα του πόσο επίκαιρη είναι η έκθεση. Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που ξεκινήσαμε. Τέλος πάντων, ε, όταν μιλάμε για συγκεκριμένες χώρες, ε, θέλουμε τρέχοντα παραδείγματα, γιατί στις χώρες υπάρχουν εξελίξεις που μετά δεν αντικατοπτρίζουν την εικόνα που δίνει η έκθεση. Εμείς ως πράσινοι βλέπουμε ότι πάντοτε η συζήτηση κολλάει σε θέματα όπως τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, ε, σεξουαλική και αναπαραγωγικά δικαιώματα, Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη. Στη, στα πλαίσια της Επιτροπής μας, είπαμε και στο διευρυμένο Προεδρείο, ότι αν πηγαίναμε στη Γενέβη, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχουν και αυτή η μεγάλη ατζέντα, έχουν πιο ε, σύντομες εκθέσεις. Ε, έχουν μόνο ένα μήνα για να κάνουν όλη αυτή τη συζήτηση. Γενικά, για αυτές τις 860 ε, τροπολογίες, να πω ότι εμείς λιγότερο από 100 καταθέσαμε και προσπαθήσαμε να είναι το σχέδιο πολύ πιο σύντομα, όπως και να έχει όμως. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή ε, αντιμετώπιση και την γραμματεία να ευχαριστήσουμε επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βερζελίπη, Η ακροαριστερά δεν εκπροσωπείται. Η Γνάτσιο Κοράο λείπει και αυτός. Οπότε να ακολουθεί κανείς και την ομάδα του. Οπότε πρέπει να δώσω το λόγο και πάει στον κύριο Βάντερ Χολτσέρ. Να πω και εγώ δύο πράγματα. Σε σχέση με αυτά που είπαμε στην αρχή. Για το κατά πόσο είναι ευανάγνωστο. Μήπως θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κάποια έτσι αρχική ανάγνωση του Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτά που λέμε ετησίως, δηλαδή να εντοπίσουμε τέσσερις ή πέντε τάσεις και να τις κοινοποιήσουμε δημόσια. Δεν ξέρω αν κάθε χρόνο χρειάζεται να ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια που τα ξέρουμε όλοι. καρμπών το κάνουμε κάθε χρόνο. Μήπως λοιπόν θα ήταν καλύτερο αντί να τα ξαναματαλέμε κάθε χρόνο να εντοπίσουμε κάποιες τάσεις ουσίας σημαντικές δηλαδή όσον αφορά την πρόσπιση των δικαιωμάτων, τη δημοκρατία κτλ. Το θέτω σε ερώτημα. Μήπως θα ήταν πιο χρήσιμο Ω δραστηριότητα τη Επιτροπής μας. Μετά, για τον κατάλογο των χωρών που αναφέρθηκε. Κάθε χρόνο λέμε ότι δεν θα αναφέρουμε κανένα και μετά αλλάζουν τα πράγματα καθοδόν. Λέμε να μην αναφέρουμε καμιά χρόνο, κανένα, καμιά χώρα και μετά συμφωνούν άλλες ομάδες να κατονομάσουμε κάποιους. με σύντομους αλλά τελείς καταλόγους χωρών. Δεν θέλουμε να φέρουμε χώρες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιες χώρες τις ξέρουμε. Εγώ θα έλεγα αναέτος να δούμε τι έχει γίνει το σημαντικό σε κάθε περιοχή του κόσμου και να αναφέρουμε τις χώρες εκεί. Και να περιζόμαστε και στις μεγάλες τάσεις, έτσι. Στις μεγάλες κατευθύνσεις. Το λέω αυτό ως ιδέα για τη συζήτηση. Δεν λέω ότι είναι τέλεια λύση, αλλά τώρα μεταξύ μας ποιος θέλει να κάνει συζήτηση και να συζητήσει τόσες τροπολογίες με τόσες συμβαστικές προτάσεις 86 και βάλε τέλο πάντων. Ε, ας κάνουμε τουλάχιστον τα πιο σημαντικά. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βαντερπότσερ, ευχαριστώντας τον αυτόν και τους άλλους εισηγητές από τις άλλες ομάδες για τη θαυμάσια δουλειά που έκαναν και ξέρω θα έχουμε μια πολύ καλή ψηφοφορία Δευτέρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για άλλη μια φορά να επενέσω τους ε, συναδέλφους γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικά, σημαντικό ότι μεταξύ μας μπορέσαμε να συνεργαστούμε τόσο καλά. Ε, λίγο σύντομα να πω ότι ε, θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να έχουμε έναν άλλο τρόπο να προχωρούμε σε τέτοιες εκθέσεις καθώς είναι όλοι έτοιμοι να το κάνουν. Ίσως σε συνεργασία με την ε, υπηρεσία έρευνες να έχουμε μία σύνοψη βάσει τις οποίες να μπορούμε να μειώσουμε τα όσα συζητάμε στην ουσία της έκθεσης. Επίσης θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά που λέμε σήμερα να είναι ε, να ισχύουν και αύριο, να είναι ξεκάθαρο τι ε, πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεωρούμε σημαντική δέσμευση αυτό που έχει αναλάβει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, όταν δεν υπάρχει απάντηση από την Κομισιόν, είναι πρόβλημα. πως είπε και ο Πρόεδρος, δεν ξέρουμε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, άρα καλό είναι να στείλουμε μια γραπ... ένα γραπτό αίτημα στην Κομισιόν να μας κάνει μια ενημέρωση σχετικά με το τι πιστεύει για αυτή την έκθεση. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι δεν πρέπει εκ των προτέρων ούτως ή άλλως να αποφασίζουμε και να κρίνουμε κάτι, γιατί έχουμε 36 ευκαιρίες μέσα στο χρόνο βγαίνουμε μέσα από τα πλαίσια των κατεπηγόντων και να εξετάζουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση από ό,τι βλέπω, λέει ο Πρόεδρος. Η ψηφοφορία είναι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 5.30 ή κάτι τέτοιο. Σωστά. Ωραία. Τελειώσαμε. Επόμενη συνάντηση στις 28 Νοεμβρίου του 2016. Τρεις μετά μεσημβρίας Βρυξέλλες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.